Bene, colleghe, Καθίστε, συνάδελφοι. Θα ξεκινήσει η συνεδρίαση γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η μερίσια διάταξη προβλέπει κάποιες πολύ σημαντικές συναντήσεις και γι' αυτό θα ξεκινήσω με την αποδοχή της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, Συνεχίζουμε τώρα στην έγκριση, με την έγκριση. Το επόμενο θέμα είναι η έγκριση των πρακτικών για τις συνεδριάσεις της 14ης Σεπτεμβρίου. Ε, νομίζω ότι εφόσον δεν υπάρχουν αγκυρίσεις θεωρούνται δεκτές. Ξέρετε ότι στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου θα πάμε στην Ιρλανδία. Μετά από την ανακοίνωση του καταλόγου των συμμετεχόντων και εχουσών, αυτό αποφασίστηκε τον μήνα Ιούλιο, μας ενημέρωσε η γραμματεία ότι τέσσερα μέλη δεν είναι σε θέση να πάνε και γι' αυτό θα Θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι θα πάνε 7 μέλη, 5 από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένας Ιρλανδός συνάδελφος και ένας πρόεδρος επιτροπής. Λοιπόν, περνάμε τώρα στα σημαντικά σημεία της ημερησίας διάταξης, το 4, Έχουμε μαζί μας την κυρία Άζα Ρέγνερ, την ε, Σουηδή Υπουργό για την παιδική ηλικία, την τρίτη ηλικία και την ισότητα των φύλων. Είμαστε ιδιαίτερος ευτυχείς που είστε μαζί μας κυρία Ρέγνερ. Όπως έλεγα λίγο πριν θα μας παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στη Σουηδία. είναι όπως λέγει η ίδια υπουργό μιας φεμινιστικής κυβέρνησης υπάρχει ειδική στήριξη στις πιο ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες και υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τη διασφάλιση και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Εγώ σαν Ιταλίδα με πολύ ε, ενδιαφέρον θα σας ακούσω γιατί στη δική μου χώρα δυστυχώς έχουμε πάρα μα πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Μας ενδιαφέρει να δούμε τι έχει γίνει στις κοινωνίες όπου έχει εφαρμοστεί πλήρως και άμεσα η ισότητα των φύλων. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στην Υπουργό η οποία θα μας παρουσιάσει κάποιες σημαντικές καινοτομίες και μετά θα δώσω το λόγο στις συναδέλφισες και συναδέλφους που θα ήθελα να θέσουν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Θα ομιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στη σημερινή συνεδρίαση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε πραγματικά κάποιες ε, κοινέ ευκαιρίες ε, αλλά και κοινέ ευθύνες για την πρόθεση των ζητημάτων ε, ίσων ευκαιριών των διοφύλων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για τη δήλωση που έκανε για την ανάγκη ύπαρξης μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για την ισότητα των δύο φύλων. Είναι πολύ μεγάλες οι προκλήσεις της σημερινής εποχής στην οποία ζούμε και τίθενται ζητήματα μεγάλα ερωτηματικά για όλους και υπάρχουν ε, Υπάρχει μια ανάγκη δράση ε, για όλου, ε, για καθέναν από εμά ξεχωριστά και για το σύνολο τη κοινωνία. Έχουμε ένοπλε σειράξει ε, γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε διαπιστώσει μια ανάγκη εκδημοκρατισμού σε πολλές χώρες. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες δημογραφικές προκλήσεις. Και ξέρουμε ότι πολλοί από αυτούς, ε, τους πρόσφυγες ε, που διωγμένοι έρχονται στην Ευρώπη, ελπίζουν ότι θα έρθουν σε χώρες όπου γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και όπου υπάρχουν αυτονόητες ε, ανθρώπινες αξίες και μία από αυτές τις αξίες είναι και η ισότητα των δύο φύλων που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο. Νομίζω ότι μπορούμε να νιώθουμε υπερήφανοι διότι στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση ε, έχει κατοχυρωθεί η ισότητα στη χάρτα των θυμελωδών δικαιωμάτων ε, και οι οργανώσεις ε, των προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών όπου έχουν αγωνιστεί και πάρα πολλοί άντρες στο πλευρό μας και ήθελα να το τονίσω ε, ανέλαβαν πολύ αποφασιστική δράση ε, και εργάστηκαν σκληρά ούτω ώστε να κατοχυρωθεί αυτή η αξία στη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και γι' αυτό θεωρώ ότι και στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει μια κοινή πολιτική για την ισότητα των δύο φυλών και να διαδραματίζει καταλητικό ρόλο σε αυτά τα ζητήματα. Το λέω ήδη στην αρχή της παρέμβασής μου για το θεωρώ σημαντικό, αλλά θα επανέλθω στη συνέχεια. Τώρα, στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, όμως υπάρχουν και πολλοί τομείς όπου ε, χρειάζεται ε, περισσότερη πρόοδος, όπως ε, διαπιστώθηκε και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Αρμόδιο για τα θέματα ισότητας των δύο φύλων. Εγώ με την ιδιότητα της Υπουργού στη Σουηδία και να η Ρίστον Παρόδο είναι η πρώτη φεμινιστική κατά τη γνώμη μου ε, κυβέρνηση στη Σουηδία και έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης 3 Οκτωβρίου πέρσι ήταν και ο Πρωθυπουργό τότε χρησιμοποίησε αυτό τον επιθετικό προσδιορισμό είπε ότι είναι φεμινιστική η κυβέρνηση. Ε, η νέα κυβέρνηση της Σουηδίας ε, και γι' αυτό και νιώθω ιδιαίτερη υπερηφάνεια διότι έχω να λάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο και μου δίνονται καταπληκτικές ευκαιρίες ε, όπως και καλούμε να αναλάβω πολύ συγκεκριμένες και πάρα πολύ βαριές ευθύνες. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε μια φεμινιστική κυβέρνηση και σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, διότι μια τέτοια φεμινιστική κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει ότι αναδεικνύει το θέμα σε προτεραιότητα, ότι διοχετεύει τα πετούμενα κονδύλια σε αυτά τα ζητήματα, ούτω ώστε να μειωθούν οι ανισότητες, ε, να προωθηθεί η ισότητα των δύο φίλων ε, και να ε, χειραφετηθούν ακόμη περισσότερο τα νεαρά κορίτσια. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν και φαινόμενα όπως οι κακές σχολικές επιδόσεις των νεαρών αγοριών. και χρειάζεται λοιπόν να διοικητεύουμε και την προσοχή μας και τα κονδύλια μας και σε άλλους τομεί όπως στην βοήθεια, στην υποστήριξη που μπορούμε να προσφέρουμε σε, στα γόρια. Κάτι άλλο που επίσης είναι σημαντικό για μας ε, είναι να δείξουμε ότι αλλάζει ολόκληρη η κοινωνία με τις εξελίξεις που σημειώνται στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσει η πολιτική ως ως δύναμη για να επέλθουν σημαντικές αλλαγές ολόκληρη την κοινωνία. Αναδεικνύοντας λοιπόν το θέμα σε προτεραιότητα, θεωρούμε ότι θα οδηγηθούμε ε, σε στρατηγική σημασία σε πρόοδο σε όλα τα ζητήματα στην ε, αγορά εργασίας, αύξηση της απασχολησιμότητας, ε, χρήση των κονδυλίων για να καλύψουμε το κενό που υπάρχει. Ξέρουμε ότι είναι μεγαλύτερο το, το ποσοστό των ε, πτυχιούχων στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια δεν δίνονται αντίστοιχα επιδόματα στους δύο γονείς ε, και μην ξεχνάμε ότι ε, υπήρξε τα τελευταία χρόνια μεγάλη αύξηση στις συντάξεις ε, των ε, αντρών ενώ δεν έχει σημειωθεί αντίστοιχη αύξηση στις γυναίκες. Υπάρχουν μεγάλες ανισότητες και αυτό που επιθυμούμε είναι ισότιμα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς το μέλλον και να δώσουμε τη σημασία που πρέπει στα σημαντικά ζητήματα. Λοιπόν, ε, η πολιτική ε, ισότητα των δύο φύλων δεν είναι ε, μια χάρη που κάνουμε στις γυναίκες, είναι προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας. Εγώ νομίζω ότι η πολιτική ισότητα των δύο φυλών απάντησε πολλά από τα σημερινά προβλήματα τη κοινωνία. Θεωρώ επίση ότι πρέπει να συμμετάσχουν εσύ το ισότιμα και οι άντρε θα πρέπει να εργάζονται στο πλευρό μα και να διαπιστώσουμε και να αποφασίσουμε ποια είναι η ευθύνη που φέρουν οι άντρε Δεν έχουν μεγαλύτερη ευθύνη σε σχέση με τις γυναίκες, όμως έχουν εξίσου μεγάλη ευθύνη και ε, βλέπουμε ότι στις περισσότερες χώρες έχουν αναλάβει την ευθύνη οι γυναίκες. Ε, ε, θα θέλαμε να μοιραστούν τις φιλοδοξίες μας οι άντρες, να εισακουστεί η δική τους η άποψη αλλά και να συμβάλλουν στην επίτευξη της προόδου. Νομίζω ότι αυτό θα είναι υποφελές όχι μόνο για τα κορίτσια και για τις νέες γυναίκες αλλά και για τα αγόρια, για τους άντρες και για το σύνολο της κοινωνίας όπως σας έλεγα. Έχουμε την εκστρατεία του ΟΗΕ, he 4 και βλέπουμε ότι τονίζεται ήδη στον ΟΗΕ η σημασία ε, του αντρικού ρόλου στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και ε, αυτό ήδη παρατηρείται στη δουλειά του ΟΗΕ για την ε, Σουηδική κυβέρνηση και συγκεκριμένα για τις εξωτερικέ υποθέσεις αλλά και στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αναδείξει το θέμα σε προτεραιότητα και έχουμε πέντε συγκεκριμένου τομεί όπου θα έπρεπε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας ε, περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας ε, μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας μείωση του μισθολογικού χάσματος ανάμεσα στα δύο φύλλα αύξηση τη ισότητας των δύο φύλων στη διαδικασία λήψη αποφάσεων καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και συμπερίληψη του ζητήματος ε, στην κατάρτιση της εσωτερικής αλλά και της εξωτερικής πολιτικής της Σουηδίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως χρηματική κυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, ε, επικεντρώνουμε την προσοχή μας αυτά ακριβώς τα ζητήματα. Φυσικά έχει σημειωθεί πάρα πολύ σημαντική πρόοδος ε, σε σχέση με άλλες χώρες αλλά και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ε, πρωτοπόροι, διότι έχουμε μικρότερε εμισθολογικέ ανισότητε, μικρότερη διαφορά στον αριθμό των γυναικών που είναι στην αγορά εργασία. Όμω δεν επαναπαυόμαστε ε, στι δάφνε μα. Για του μισθού, παραδείγματο χάρη, στη Σουηδία καθορίζονται από την ίδια την αγορά εργασία και όχι από τη Σουηδική κυβέρνηση, όμω ασκούμε πίεση με άλλου τρόπου για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα για την βία κατά των γυναικών. Γίνονται πάρα πολλά πάρα πολλές προσπάθειες ε, να προστατεύσουμε τις εκτεθειμένες ε, γυναίκες ε, και τα παιδιά. Λέω παιδιά διότι μπορεί να είναι αγόρια ή κορίτσια και... Επίσης έχουμε εφημερίες με αρκετούς οικονομικούς πόρους, ούτως ώστε να υπάρξει μια ικανοποιητική υποδοχή για τις γυναίκες που έχουν υποστεί Έχουμε μια από τις πιο πρωτοποριακές νομοθεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την σεξουαλική βία κατά των γυναικών το πρόβλημα δεν είναι όμως μόνο ε, η ε, βία και παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα 15-20 τελευταία χρόνια παραμένει αυτό το φαινόμενο και μπορώ να πω σε ορισμένε ε, περιπτώσεις έχει επιδεινωθεί. το θέμα είναι η πρόληψη της βίας, ούτως ώστε να μην συμβεί ο βιασμός, να μην γίνει η σεξουαλική επίθεση κατά των γυναικών, να είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ζητημάτων με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί μια φεμινιστική κυβέρνηση. Στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση σίγουρα δεν θα έχουμε επιλύσει όλα αυτά τα ζητήματα, θα εκκρεμούν ακόμη πολλά θέματα, όμως θέλουμε να δείξουμε ότι έχουμε λάβει σωστέ αποφάσει ότι έχουμε ιεραρχήσει τις προτεραιότητε μας και έχουμε ε, επαρκείς ε, ε, πόρους για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση που έχουμε προκρίνει για το, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτά τα ζητήματα, επειδή ξέρουμε πόσο μεγάλη βαρύτητα έχουν αυτά τα θέματα σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούμε ότι μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την ισότητα των δύο φύλων έχει ιδιαίτερη σημασία για να υποστηρίξουμε τις εξελίξεις, να προωθήσουμε τις εξελίξεις που σημειώνονται σε κράτη-μέλη και για να δίνει το παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην παγκόσμια σκηνή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, μακρόπνο και με στρατηγικό τρόπο να εκπονούμε τις προτεραιότητές μας στον τομέα της ισότητα των δύο φύλων. Εάν δούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί έχουμε και πολύ καλά στατιστικά στοιχεία από το αρμόδιο Ευρωπαϊκό Οργανισμό, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε χαμηλότερες αμοιβέ, χαμηλότερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας ε, και κατάρτιση. Ε, υπάρχουν λήψεις στις ε, δομές ε, ε, όπως η βρεφονιπιακή σταθμή, παραδείγματος χάρη, τα νηπιαγωγεία, ε, και ε, διαπιστώνουμε τα προβλήματα των γυναικών ξεκινούν πολύ συχνά από αυτό, διότι πρέπει να φροντίζουν τα παιδιά τους ηλικιωμένους, διότι λείπουν αυτές οι απαιτούμενες δομές. Και Ε, δεν, έχουν, ε, δεν έχουμε προς το παρόν ε, ικανοποιητικές εξελίξεις σε πολλά κράτη-μέλη. Χαμηλότατη συμμετοχή επίσης στα κοινοβούλια σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, να έχουν καλύτερη κατάρτιση και εκπαίδευση οι γυναίκες, να καταπολεμηθεί η ε, σεξουαλική βία κατά των γυναικών και το καθεξής. Τα ίδια ζητήματα τίθενται δηλαδή και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο να ε, παίξει στη, σε παγκόσμια κλίμακα για την υπεράσπιση των γυναικών, για την καταπολέμηση των διακρίσεων ε, ε, βάρος τους ε, για την καταπολέμηση της φτώχειας ε, των γυναικών. Η ισότητα των δύο φύλων είναι μια βασική προϋπόθεση ούτως ή άλλως για να επιτύχουμε την βιώσιμη ανάπτυξη, την ασφάλεια και την ειρήνη στον κόσμο τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών θα πρέπει να εξακολουθήσουν να συνιστούν προτεραιότητα στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και να καθοδηγούμε τη δράση μας προς αυτή την κατεύθυνση μετά και την έγκριση των νέων στόχων της ε, χιλιετίας. Ε, ε, στη, υπήρξε και μια διάσκεψη στην Λατινική Αμερική ε, για την, τα δικαιώματα των γυναικών και εκεί είδα επί τόπου πόσο μεγάλο βάρος έχει η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον υπόλοιπο κόσμο. είναι πάρα πολύ σημαντική η δράση μας και εκεί πέρα βλέπουμε πόσο, πόσο ειδικό βάρος έχουν τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθεί στις εξωτερικές τη για την πρόθεση αυτών των ζητημάτων. Η Σουηδία για την ασφάλεια και τις εξωτερικές ε, υποθέσεις ε, έχει μια ιδιαίτερη υπηρεσία ούτως ώστε ε, στο υψηλότερο επίπεδο να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις στον ΟΗΕ όπως θα ψηφίσουμε τα 1325 και 1820 ε, και θέλουμε να ε, συσταθεί και η ειδική επιτροπή για αυτά τα ζητήματα στον ΟΗΕ. Θα θέλαμε λοιπόν να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσουμε και αυτή την προτεραιότητα, διότι είναι πολύ, σημαντικά, πολύ σημαντικές οι δράσεις που αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΟΗΕ. Εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να διαπιστώσω για ποιο λόγο Ποια είναι η βαθύτερη αιτία που μας ε, ε, αποτρέπει από την υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για την ισότητα των δύο φύλων, διότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια απάντηση στα σημερινά μας προβλήματα. Ε, στην εποχή που ζούμε, αν δεν το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος θα το κάνει. Τι κάνει λοιπόν μια φεμινιστική κυβέρνηση. Πώς περνάμε από τα λόγια στη δράση. Αλλά πρώτα απ' όλα όντως είναι σημαντικά τα λόγια. Είναι σημαντικός ο διάλογος, ο διάλογος για τα ζητήματα αυτά. Ε, τα τελευταία 100 χρόνια γίνεται, συνεχίζεται αυτός ο διάλογος, πόσο μπορούμε να ενισχύσουμε το ρόλο των γυναικών, να προωθήσουμε τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών. Δικαίωμα ψήφου δεν θα είχαμε αν δεν υπήρχε αυτός ο διάλογος ακόμη. Ε, Βεβαίω δεν είναι μόνο σημαντικά τα λόγια αλλά και οι πράξεις και η ε, στρατηγική δράση. Πρέπει να στοχοθετούμε και να υλοποιούμε. Ε, έχουμε μια μακρά παράδοση στη Σουηδία για την ενσωμάτωση αυτού του ζητήματος ε, ε στους όλους τους τομείς. Στο Πεκίνο, όπως ξέρετε, το 1995 έγινε μια συγκεκριμένη πρόταση για να ενσωματωθεί η διάσταση ισότητας των δύο φύλων σε όλα τα έγγραφα εργασίας. Τότε αρχίσαμε κι εμείς και συνεχίσαμε έκτοτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το mainstreaming, όντως, ε, και με την φεμινιστική κυβέρνηση εντατικοποιήσαμε και την εργασία στον τομέα αυτό και αυξήσαμε και τον αριθμό των υπηρεσιών που ε, με στρατηγικό τρόπο ε, ασχολούνται με την ε, συμπερίληψη της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων σε όλους τους τομείς δράσης της κυβέρνησης. Πού πρέπει να μας οδηγήσει όμως αυτό το mainstreaming. Είναι επίσης ε, σημαντικό να συνδυαστεί με άλλα εργαλεία για να ξέρουμε ποιος ακριβώς ε, φέρει την ευθύνη. Καλό είναι να εργαζόμαστε όλοι για τον ίδιο στόχο. Όμως κάποιος πρέπει να λογοδοτεί, κάποιος πρέπει να έχει την πρωταρχική ευθύνη. Στη φεμινιστική μας ε, κυβέρνηση θέλουμε λοιπόν ε, να ε, ολοκληρωθεί και η εργασία μας στον τομέα της κατάρτισης ε, του προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των κονδυλίων για τα ζητήματα αυτά. Τις ερχόμενες εβδομάδες θα αποφασιστεί, θα εγκριθεί το σχέδιο προϋπολογισμού εξάλλου στη Σουηδία και θα θέλαμε σε εθνικό επίπεδο να προωθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση τον προϋπολογισμό των κονδυλίων. Τι εννοώ. Πρέπει να υπάρξει μία εμπεριστατωμένη ανάλυση σε σχέση με το πώς θα γίνει η κατανομή των των κονδυλίων και με το ποιο τρόπο θα επηρεάσει αυτό τι εργασίε μα στον τομέα τη προώθησης τη ισότητα των δύο φύλων, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε αποτελέσματα συγκεκριμένα, να αυξάνεται η ισότητα των δύο φύλων. Έγιναν σοβαρές προσπάθειες για να το καταφέρουμε αυτό και ε, στις επόμενες εβδομάδες θα γίνουν ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις ε, για να διαπιστώσουμε ακριβώς πώς μπορεί να αποτυπωθεί αυτό στο σχέδιο προϋπολογισμού και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε την περαιτέρω στον τομέα. Υπάρχουν, ξέρετε, διαφορετικά, διαφορετικοί μορφότυποι για να προϋπολογίσουμε κατάλληλα τα κονδύλια και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο αριθμοί, επηρεάζεται η καθημερινή ζωή των γυναικών, των κοριτσιών, των ε, αγοριών, των αντρών και ολόκληρης της κοινωνίας. Ε, για να ξέρουμε λοιπόν ε, προς τα που πορευόμαστε θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους στόχους και να αντιμετωπίζουμε τους τομείς προτεραιότητες και τα εκκρεμή ζητήματα ούτως ώστε επιτόπου να αναλάβουμε συγκεκριμένη και αποτελεσματική δράση το να ε, επιτύχουμε το mainstream χωρίς να έχουμε χάρτη πορείας δεν μας βοηθάει και πάρα πολύ. Πρέπει να έχουμε απτά αποτελέσματα εσχάτως. δημοσιεύθηκε και μία έκθεση για τις εργασίες ε, της ε, κυβέρνησης, φεμινιστικής κυβέρνησης για αυτά τα ζητήματα. Από το ελεγκτικό μας συνέδριο και διαπιστώθηκε ότι όντω έχουν επενδυθεί κονδύλια και τον περασμένο χρόνο έχουν γίνει βήματα που χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Έχουν δρομολογηθεί πολύ σημαντικά προγράμματα, όμως δεν λείπει η σωστή κατεύθυνση, δεν υπάρχει καταμέτρηση των αποτελεσμάτων και δεν είναι σαφής η εικόνα τελικά ε, των αποτελεσμάτων. Αυτό θα πρέπει να το αλλάξουμε για να διαπιστώνουμε αν έχει ή όχι σημειωθεί η οχι σημειωθει η Για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία ε, αυτό το ε, ζήτημα του, της κατάντια αποτίμησης της δράσης μας. Oh. Jag ser att den tid vi lever i Στη σημερινή εποχή έχουμε όχι μόνο τις μεγάλες προκλήσεις, τα μεγάλα προβλήματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθουμε, αλλά διαπιστώνουμε πως έχουμε και νέες ευκαιρίες για να προωθήσουμε την, ε, την ισότητα των δύο φύλων. Όπως σας έλεγα, με μια καλά κατερδισμένη στρατηγική μπορούμε να συμβάλλουμε στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων της κοινωνίας γενικότερα και ειδικότερα να βελτιώσουμε τη ζωή πολλών αντρών και γυναικών. Η επόμενη γενιά ίσως δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει ακριβώς γιατί χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως όταν βλέπουμε ότι άλλα υπόσχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα υπόσχονται και τα κράτη-μέλη και άλλα κάνουν τελικά. Υπάρχει μια αντιστοιχία. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν φιλοδοξίες όπως η ισότητα των δύο φιλών στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων όμως πρέπει να αποδείξουμε ότι και στην πράξη είμαστε στο πλευρό των γυναικών και των εντρών και θα αγωνιστούμε στο πλευρό τους και θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Καλό είναι να έχει σημαντικέ φιλοδοξίε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και για τη σεξουαλική βία και την αναπαραγωγική υγεία. Γιατί και πάλι θα το ξαναπώ, αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει. Η νέα αναπτυξιακή στόχη του ΟΗΕ, και θα κλείσω σε λίγο, έχουν αποφασιστεί και σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται η ισότητα των δύο φύλων, ε, οι οργανώσεις ε, προάσπισης ε, των γυναικών και των κοριτσιών που έχουν αγωνιστεί σκληρά τα τελευταία χρόνια μας βοηθούν και δίνουν το ένασμα για ανάληψη αποφασιστικότερες δράσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρώ επίσης ότι σήμερα ε, βιώνουμε μια αλλαγή ε, στον τομέα αυτό στον κόσμο. Συζητούσαμε μια γυναίκα ρόμ στην ε, Σουηδία που λέγεται Ρενάτα Φέιτσολίτς και είναι ακτιβίστρια στη, στη Στοκχόλμη και συζητούσαμε γενικότερα για τα συζητήματα ισότητας των δύο φίλων και μου μίλησε για αυτήν την ε, μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει πλήττεται από υψηλή ανεργία, ε, χαμηλότερη εκπαίδευση, ε, κακή στέγη, κακή υγειονομική περίθαλψη και συχνά οι γυναίκες είναι σε δυνότερη θέση σε σχέση με τους άντρες. Και τη ρώτησα, έχεις εσύ ένα συγκεκριμένο μήνυμα, θέλεις να περάσω ένα συγκεκριμένο μήνυμα από πλευρά σου σήμερα στην Επιτροπή των Γυναικών και μου λέει ναι θα ήθελα όταν κάποιος βλέπει ένα νεαρό κορίτσι ρομ να σκεφτεί κάποιος να μία μέλουσα μηχανικός, μία μέλουσα επιστήμων, μία ε, επιχειρηματίας, μία διευθύντρια, ένα κορίτσι στο οποίο αξίζει να επενδύσουμε Χρειαζόμαστε όλα τα κορίτσια, όλες τις γυναίκες που μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που το δικαιούνται. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ προσωπικά, ευχαριστώ και εξ ονόματος της Επιτροπής την κυρία Ρέγνερ μιας γυναίκας που δίνει αγώνα όπως όλες μας ανεξάρτητα από την πολιτική μας καταγωγή. Και εμείς δίνουμε αγώνα για όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρατε. Προσπαθούμε να κρατήσουμε το θέμα αυτό ε, σαν προτεραιότητα αυτών οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική. πρέπει στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να υπάρχει η πλευρά, το θέμα της ισότητας των ευκαιριών. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα οποία μόλις μας είπατε μας φαίνονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ε, στο πρόσωπο όλων εδώ δεν θα έχετε παρά μόνο συμμάχους Με μεγάλη χαρά βλέπουμε μία υπουργό, μία γυναίκα καταρχάς, κάτι το οποίο μας δίνει περισσότερες ελπίδες. Όπως είπαμε ο προϋπολογισμός θα λαμβάνει υπόψη του το θέμα του γένους, του φίλου συγγνώμη, Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα αμοιβών, όχι μόνο στη δική σας χώρα, αλλά και στις υπόλοιπες. Λοιπόν, οι συνάδελφοι μπορούν να θέσουν ε, ερωτήσεις. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώνασον, αν δεν κάνω λάθος, έχει προτείνει ένα νόμο ο οποίος προβλέπει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του 40% γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των σουηδικών επιχειρήσεων. Ε, πού βρίσκεται η συζήτηση για αυτό το νόμο. Πότε προβλέπετε ότι θα υιοθετηθεί. Θα ξεκινήσω με την συνάδελφο Βίμπεργκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όσα για την ενημέρωση. Δεν έρχονται και κάθε μέρα οι υπουργοί από τη Σουηδία. Δεν είναι πολύ ευχάριστο ε, για, την, ε, για τον οκροτηριασμό των σεξουαλικών ε, οργάνων των γυναικών, ιδιαίτερα ε, επίπονη μαρτυρική διαδικασία που επηρεάζει την υγεία των γυναικών μακροπρόθεσμα. Τρία εκατομμύρια γυναίκες αντιμετωπίζουν αυτό τον κίνδυνο, αυτήν την απειλή βάσει της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Πρόκειται για βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, κατάχρηση εξουσίας και η απειλή ε, ε, και απειλούνται πάρα πολλές ε, γυναίκες με καταστολή ουσιαστικά της σεξουαλικότητάς τους αυτό το φαινόμενο δεν θα έπρεπε να παρατηρείται πουθενά στον κόσμο αλλά κυρίως όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να σε ρωτήσω ξέρεις πόσα κορίτσια βρίσκονται σε ζώνες, σε, επικίνδυνες ζώνες στη Σουηδία και απειλούνται με αυτόν τον ακροτηριασμό των σεξουαλικών τους οργάνων. Έχει ξεκινήσει η δράση από το 1990 ε, και έχουν γίνει βήματα όμως ε, για την πρόληψη και την αποτροπή ε, του ακροτηριασμού. Τελικά δεν έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα και υπάρχουν επίσης άλλου κυρώσεις από τις κοινότητές τους ε, ε, ή ε, πηγαίνουν τα κορίτσια, τα στέλνουν για τις καλοκαιρινές διακοπές στη χώρα προέλευση τους για να γίνει ο των γεννητικών οργάνων όταν προσπαθούμε εμείς να τους εμποδίσουμε στη Σουηδία. Και επίσης ο αριθμός των βιασμών, έχουμε τον υψηλότερο αριθμό βιασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ντρέπομαι που το λέω και υπάρχουν ε, όχι μόνο ατομικοί αλλά και ομαδικοί βιασμοί. Τι κάνει το Υπουργείο λοιπόν για να καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο διότι δεν έχουμε ε, καθόλου καλά αποτελέσματα. Διαρκώς αυξάνει το αριθμό των βιασμών. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις εκ των Grazie. La parola alla collega Morvai. Morvai. Köszönöm szépen. Az előbb Ευχαριστώ πρόεδρε. Η συνάδελφος προηγουμένως αναφέρθηκε σε μια πρακτική, τον ακροτηριασμό των γενετήσεων δηλαδή, λέγοντας ότι έχει πολιτιστικές καταβολές. Και εσείς Υπουργέ αναφερθήκατε στον πολιτισμό ε, των Ρώμα και είπατε ότι θα θέλατε όταν κάποιοι βλέπουν μια νέα τσιγκάνα στο δρόμο να πιστεύουν ότι θα γίνει μια μελλοντική επιστήμον. Πώς αντιμετωπίζετε εσείς στη χώρα σας τις πολιτιστικές διαφορές και τι πιστεύετε για τις διακρίσεις οι οποίες ε, βασίζονται στις πολιτιστικές ε, διαφορές. Υπάρχουν πολλές μειονότητες, όχι μόνο η Ρωμά. Πρέπει να βοηθούμε λοιπόν τις μειονότητες και αν θέλουμε οι νέοι Ρώμα να αντιμετωπίζονται σαν μελλοντικοί πολιτικοί, μηχανικοί, επιχειρηματίες κτλ. Τότε θα έπρεπε να δούμε και τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν από τον πολιτισμό και τις οικογένειες αυτών των παιδιών, αυτών των κοριτσιών. Μήπως θα πρέπει οι οικογένειες να βοηθήσουν έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύ συχνά αυτές οι γυναίκες αναγκάζονται να παραμείνουν στο σπίτι, να μην πάνε στο σχολείο για να βοηθήσουν για την ανατροφή των αδελφών τους. Συνεπώς, έχω την εντύπωση ότι τα περισσότερα προβλήματα για τις Ρώμα προέρχονται από το εσωτερικό των οικογενειών τους αν θέλετε οι γυναίκες αυτές να γίνουν επιχειρηματίες και επιστήμονες θα πρέπει να δείτε τα εμπόδια τα οποία δημιουργούν οι ίδιες τους οι οικογένειες. Αναφερθήκατε με πολύ θετικό τρόπο και στο θέμα της μετανάστευσης. Ξέρετε τι εικόνες βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ή βλέπουμε στις ειδήσει Βλέπουμε ότι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν πολλοί, εκπροσωπούνται πολλές χώρες και πολιτισμοί όπου οι γυναίκες αντιμετωπίζονται ε, με βίαιο τρόπο. Ίσως να ομιλώ για θέματα δύσκολα, αλλά πρέπει να με αφήσετε να τελειώσω όπως αφήσατε την προλαλή Αν θέλετε να βάλετε χρονόμετρο, αλλά να το λέτε εξ αρχής για πόση ώρα μπορώ να μιλήσω. Δεν μου είπατε για πόση ώρα μπορώ να μιλήσω και γι' αυτό θα τελειώσω την παρουσίασή μου. Λοιπόν, κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε για την αντιμετώπιση των γυναικών από πλευράς των μεταναστών Ε, πώς συμπεριφέρονται στις γυναίκες τους και στα παιδιά τους όταν ε, ε, επιλέγουν το ποιοι θα ανέβουν στα τρένα λοιπά. Βέβαια με αυτά τα οποία λέω σας δημιουργώ πανικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει τι κάνετε για να παρεμποδίσετε τους μουσουλμάνους αυτούς μετανάστες να βιοπραγούν εις βάρος των παιδιών τους. Ηρεμήστε συνάδελφε λέει η πρόεδρος. Όχι θα με αφήσετε να τελειώσω λέει η ομιλήτρια. Η κυρία Μόρφα είμαι μέλος του κοινοβουλίου όπως εσείς και περιμένω απαντήσεις. Συνάδελφε κοιτάξτε. Όταν σας λέω παρακαλώ περιορίστε το χρόνο σας, αυτό είναι γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Εγώ δεν θέλω να είμαι δικτάτορ εδώ και να επιβάλλω διάφορους χρόνους στον καθένα. Ε, ίσως είσαστε στο κοινοβούλιο πιο πολύ από μένα και ξέρετε ότι δεν πρέπει να μελάτε για πάνω από 5 λεπτά, 5 ή 7 λεπτά. Λοιπόν, εάν κάποιος όμως μιλάει περισσότερο, έστω και ένα 1,5 λεπτό, εγώ απλά χτυπώ το σφυράκι μου εδώ για να δώσουμε ακριβώς στην Υπουργό το χρόνο ε, απάντησης και γενικά αναστατώσατε τη συζήτηση και αυτό δεν δημιουργεί καλές συνθήκες για την απάντηση. Λοιπόν, η επόμενη συνάδελφος είναι η κυρία Χόνεμπολ. Όχι, η κυρία Μπιόρκ έχει το λόγο, λάθος έκανα. Θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Υπουργό διότι συνήθω είμαστε αρκετά ήρεμε στην Επιτροπή, ούτε βάραμε τραπέζια, ούτε τίποτα. Δεν θέλω όμω να έχετε σε καμία περίπτωση την εντύπωση ότι αφήνουμε του ρατσιστέ να κάνουν κουμάντο στι συνεδριάσει. Συνήθω δεν ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των γυναικών. Και αυτό είναι τελείω άκομψο. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω τώρα τη μητρική μου γλώσσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Ξέρω ότι έχει αναλάβει σοβαρότατη δέσμευση για την ισότητα των δύο φύλων, για την καταπολέμηση της βίας, ε, για την πρόθεση των ε, σεξουαλικών και αναπαραγωγικών ε, δικαιωμάτων. Δεν είμαστε από την ίδια πολιτική οικογένεια, αλλά φυσικά όλοι αναπνέουμε, είναι, μια, είναι φρέσκος αέρας για μας, αναπνέουμε όλοι καλύτερα από τότε που ορκίστηκε αυτή η φεμινιστική κυβέρνηση Ζητώ συγγνώμη που μπορεί να ακούγεται αυτό που θα πω όσο ότι εσύ έχεις μια απόλυτη επιρροή στο Συμβούλιο. Δεν εννοώ αυτό, αλλά τέλος πάντων θα ήθελα να ξέρω τι μπορείς να κάνεις. Ε, μας απασχολούν ε, πάρα πολλά από τα ζητήματα που ανέφερες ε, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το εξή. το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δική της πολιτική για την ισότητα των διοφύλων του. Στο Συμβούλιο έχουμε τη δήλωση του τρίου των Προεδριών και θεωρούμε ότι εδώ στην Επιτροπή των Γυναικών ότι αρκούν αυτά τα λόγια και θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη η στόχη αν θέλουμε πραγματικά να γίνει κάτι. Δεν φτάνει αυτό που κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο, δεν φτάνει αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό συνασπισμό για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών. Αυτό χρειάζεται το τρίο των Προεδριών, μεγαλύτερη, σημαντικότερη δέσμευση. Τώρα πώ εσεί μπορείτε να μας βοηθήσετε στο Συμβούλιο Συμβούλιο ε, για να επιτύχουμε τους στόχους μας εδώ στην Επιτροπή των ε, Γυναικών. Αποσύρθηκε η πρόταση για την ε, άδεια μητρότητας. Έχει επανέλθει στο Συμβούλιο. Τι θα γίνει με αυτό, τι μπορείτε να κάνετε για να μας βοηθήσετε γιατί το νέο νομοσχέδιο τα ξέρεις όπως και εγώ αλλά ήθελα να μιλήσω για το εμπόριο γυναικών και για την πορνεία. Ε, διακόπτη η πρόεδρος την κυρία Μπιόρκ. Η κυρία Χάνιμπολ τώρα. Μη με αναγκάζετε να σας θυμίζω το χρόνο, γι' αυτό παρακαλώ ε, απευθύνω έκκληση στην κοινή λογική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ που ήρθατε εδώ σήμερα. Θα είμαι πολύ σύντομη, διότι θα ήθελα να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη ομιλήτρια, η πορνεία δηλαδή, και πώς θα μειώσουμε τη ζήτηση στην πορνεία. Όπως ξέρετε, πέρυσι το Κοινοβούλιο ψήφισε μια έκθεση η οποία εγκρίνει στην ουσία το σουηδικό μοντέλο. Και ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη για αυτήν εδώ την Επιτροπή. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να πάμε ακόμα παραπέρα και θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό σε όλη την επικράτεια της Ένωσης διότι υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα πορνείας όπως ξέρετε. Υπάρχουν και ορισμένες χώρες στις οποίες η πορνεία είναι νόμιμη. Πρέπει όμως νομίζω να καταλήξουμε σε μια κοινή ευρωπαϊκή οπτική γωνία ακόμα και αν η νομοθεσία είναι στο χέρι των κρατών μελών διότι η πορνεία συνεπάγεται και τη διακίνηση ανθρώπων κάτι σύνηθε στην επικράτεια της Ένωσης ε, θα ήθελα λοιπόν εγώ να, να ακούσω τις ε, σκέψεις σας για το πώς ε, μπορούμε να εφαρμόσουμε το σουηδικό μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα πείσουμε το Συμβούλιο να το ακολουθήσει. η κυρία Πόστ. Θυμίζω ότι η Υπουργό θα πρέπει να φύγει στις 4. Ελπίζω να μπορέσει να μείνει λίγο παραπάνω. Η κυρία Πόστ έχει το λόγο. Όχι, για το αποσύρω δεν θέλω να κάνω ε, ερωτήσεις. Ε, ζήτησα το λόγο διότι είναι ακροδεξιές οι δηλώσεις που ακούσαμε εδώ από τη συναδελφή και ε, με αυτό το φανατισμό το ρατσιστικό που έχει δεν θα έπρεπε καν να της επιτρέπεται να επεμβαίνει. Αλλά μόνο γι' αυτό ζήτησα το λόγο. Ήθελα να διαμαρτυρηθώ εντόνως. Rodríguez. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση. Έχω δύο πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα για σας. Πρώτον, με ποιο τρόπο καταπολεμάται ένα στερεότυπο το οποίο όμως διατηρείται από την ίδια την κυβέρνηση, ο Υφυπουργός, ο αρμοδίος Υφυπουργός της ε, Πορτογαλίας είπε ότι πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά να πληρώνουν τους λογαριασμούς και να καθαρίζουν το σπίτι οι γυναίκες. Ε, οπότε θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει ε, πρόγραμμα δράσης στη Σουηδία για τις ε, γυναίκες που έρχονται από τη Μεσόγειο. Πώς μπορεί δηλαδή να επικρατήσει αυτή η σουηδική λογική και στις υπόλοιπες χώρες, κυρίως στις νότιες χώρες. Έτσι πρέπει να τίθενται οι ερωτήσεις. Η Υπουργός Ρέγνερ έχει το λόγο. Thank you very much. Um, okay. Thank you for your interest in, in English. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δείξατε. Πρέπει στις 4 να πάω σε άλλη συνεδρίαση, γι' αυτό λοιπόν συγχωρήστε μου την ε, σύντομη απάντηση. Θα χαρώ πολύ να συνεχίσουμε την επαφή μας και να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα, όπως για παράδειγμα την ε, διαφορετική νομοθεσία, τη δική μας νομοθεσία στη Σουηδία για την ε, πορνεία. Αυτό σίγουρα μπορούμε να το συζητήσουμε περισσότερο. Και είναι μάλιστα ένα θέμα το οποίο αλλάζει συνεχώς. Εάν θέλετε λοιπόν είμαι στη διάθεσή σας. Τώρα, ε, σχετικά με τον ε, συνάδελφο μου Υπουργό Δικαιοσύνη που είναι επίσης και Υπουργό Μετανάστευσης και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Αναφέρεται στις κυβερνητικές δηλώσεις ότι εάν εάν οι συγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείε δεν έχουν το 40%, 40 ε, γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια μέχρι το 2016, τότε θα νομοθετήσουμε για αυτό. Φαίνεται πως ε, μέχρι τώρα το ποσοστό αυτό έχει φτάσει στο 30%. Και ελπίζω πως οι ίδιες οι εταιρείες θα καταφέρουν μόνες τους να εκπληρώσουν το στόχο του 40% του χρόνου. Εάν δεν συμβεί όμως κάτι τέτοιο, τότε φυσικά θα προτείνουμε νομοθεσία στο χώρο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντλούμε ανθρώπινο δυναμικό και από άντρες και από γυναίκες. Και φυσικά είναι επίσης ε, αλήθεια ότι λαμβάνονται πολλές αποφάσεις που επηρεάζουν την κοινωνία σε τέτοια επίπεδα διοικητικών συμβουλίων. Ε, λαμβάνονται αποφάσεις που θα επηρεάσουν τα επόμενα 10-15 χρόνια μιας κοινωνίας. Βέβαια, να σας πω πως δεν έχουμε κάποιες ποσοστώσεις ούτε στην πολιτική ούτε κάπου αλλού. Θα είναι λοιπόν πρώτη φορά που θα ε, ασχοληθούμε επίσημα με κάτι τέτοιο και ελπίζω λοιπόν αυτό το 40% γυναίκες να ε, έρθει μόνο του και να μην χρειαστεί εμεί να νομοθετήσουμε. Όσον αφορά για τον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων, εδώ και χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό είναι και άλλωστε στα πλαίσια της πλατφόρμας του Πεκίνου και του Καΐρου. Υπάρχει νομοθεσία στη Σουηδία γι' αυτό. Ετέθησε ισχύ πέρυσι. Βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να αφήνουμε από τα μάτια μας. Πρέπει συνέχεια να συζητούμε και να υπάρχει διαρκής ενημέρωση και φυσικά κατάλληλη νομοθεσία. Σχετικά με τους βιασμούς τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε πως μειώνεται η βία κατά των γυναικών, όμως νομίζω πως ε, δεν παρατηρείται τάση για αύξηση στους ομαδικούς βιασμούς. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία. Βέβαια, Ο βιασμός είναι ένα απεχθές έγκλημα κατά μιας γυναίκας. Γι' αυτό λοιπόν και αυτή τη στιγμή αναθεωρείται η νομοθεσία σχετικά με τα σεξουαλικά εγκλήματα και τα σεξουαλικά δικήματα. Ε, τώρα, όσον αφορά την ένταξη, φυσικά και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντική ένταξη των προσφύγων που φτάνουν στη Σουηδία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας και είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι μπορούμε να υποδεχτούμε πρόσφυγες οι οποίοι ε, φεύγουν από εμπόλεμες ε, περιοχές, φεύγουν από χώρες τις οποίες επικρατούν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, ε, από τη Συρία για παράδειγμα. Θεωρούμε πως είναι καθήκον μας να βοηθήσουμε και είμαστε περήφανοι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό φυσικά συνεπάγεται ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε ε, άνδρες και γυναίκες και παιδιά στη χώρα μας. Ε, περίπου πάνω από τους μισούς πρόσφυγες είναι παιδιά. Και βλέπουμε ότι καθώς αυξάνονται οι πρόσφυγες, αυξάνεται και η ανάγκη για ένταξή τους. Πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε για τη στέγασή τους, για την ένταξη στην αγορά εργασίας, για την παιδεία και ούτω καθεξής. Σχετικά με τις γυναίκες τώρα. Πράγματι, η συμμετοχή στην αγορά των γυναικών είναι χαμηλότερη από εκείνη των ε, ανδρών, σε συγκρίσιμες ομάδες. Μπορούμε όμως να πούμε επίσης ότι αυξάνονται τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών περισσότερο από εκείνα των ανδρών. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε γιατί. Να ε, δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πιστεύω και ελπίζω πως οι γυναίκες και οι άνδρες θα βλέπουν τη Σουηδία ως μια χώρα στην οποία θα θέλουν να πάνε, ως μια χώρα στην οποία επικρατεί ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και πως ε, και οι άνδρες και οι γυναίκες θα θεωρούν ότι αυτές είναι σωστές, καλές αξίες. Και πέραν από τις άλλες μου ιδιότητες είμαι και υπουργό αρμόδια για τα δικαιώματα των παιδιών και στα καθήκοντά μου είναι και η αλλαγή του δημογραφικού προβλήματος. Αυτή τη στιγμή η παροχή φροντίδας στους ηλικιωμένους είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Περίπου 5% του εργατικού δυναμικού στη Σουηδία ασχολείται με την φροντίδα ηλικιωμένων. Είναι θέσεις εργασίας που χρηματοδοτούνται από το κράτος κατά μεγάλο ποσοστό. Αυτός ο χώρος είναι γυναικοκρατούμενος θα έλεγα. Ε, θα ήθελα να υπήρχαν περισσότεροι άνδρες ε, που να εργάζονται στο χώρο αυτό. Σίγουρα θα χρειαστούμε περισσότερους φροντιστέ ηλικιωμένων στο μέλλον. Ωστόσο πρέπει να πω ότι εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι νέοι Σουηδοί, οι πρόσφυγες, άλλοι ε, μετανάστες που έφτασαν στη χώρα μας. Εάν δεν είχε αυξηθεί λοιπόν ε, ο πληθυσμός με αυτούς τους νέους Σουηδούς, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρναμε στο μέλλον και ε, πώς θα καταφέρναμε να χρηματοδοτήσουμε το σύστημα αυτό με τα χρήματα των φορολογούμενων και πώς θα είχαμε αυτό το εργατικό δυναμικό να εργάζεται στον χώρο αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια μεγαλύτερη φορολογική βάση την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη φροντίδα ηλικιωμένων. Εάν δεν υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι άντρες και γυναίκες δεν θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ούτε την ε, παιδική μέρημνα ούτε την ε, φροντίδα των ηλικιωμένων. Είμαστε λοιπόν χαρούμενοι για το γεγονός ότι έχουμε αύξηση του πληθυσμού μας όσον αφορά την ισότητα μεταξύ των φίλων. Θα ήθελα να πω ότι μέχρι τώρα δεν έχω επίγνωση καμίας ε, χώρας όπου δεν έπαιξε ρόλο η πολιτική. Η πολιτική άλλαξε το κατεστημένο οι πολιτικές ιδέες, η πολιτική θέληση και το γυναικείο κίνημα. Άλλαξε λοιπόν τα δεδομένα και όχι οι ατομικές ε, προσπάθειες τόσο πολύ. Και πιστεύω πως χρειάζεται λοιπόν αυτή η πολιτική βούληση για να επιτύχουμε την ισότητα. σχετικά με το Συμβούλιο τώρα. Φυσικά και πιστεύω πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα σε θέματα ισότητας. Και κυρία Μπιόρκ, με τα χαρά να το συζητήσω περισσότερο μαζί σας. Πιστεύω, όπως είπα, ότι είναι αναγκαίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εργαστεί περισσότερο σε αυτόν τον τομέα και πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων. Γι' αυτό λοιπόν με τα χαράς, όπως σας είπα, να συζητήσουμε και διμερώς πάνω σε αυτό. Επίσης, σχετικά με την οδηγία για την ε, άδεια μητρότητας, η θέση της κυβέρνησής μας ήταν να συμπεριλαμβάνονται και οι μητέρες και οι πατέρες στην γονική άδεια. Γι' αυτό λοιπόν και την ονομάσαμε γονική άδεια και όχι άδεια μητρότητας. Και πάλι θα χαρώ πολύ να το συζητήσω μαζί σας και να πω πως ε, χαίρομαι ιδιαίτερα με το ότι συζητούμε αυτό το θέμα. Η γονική άδεια στη Σουηδία αυξήθηκε και αποφασίσαμε μάλιστα να την κάνουμε υποχρεωτική και για τους δύο γονείς. Από τους 12 μήνες λοιπόν γονικής άδειας πρέπει τουλάχιστον οι δύο ε, να χρησιμοποιηθούν από τον ένα γονιό. Τώρα τους αυξήσαμε στους 3 μήνες, στους 12. Όταν λοιπόν μια οικογένεια κάνει παιδί, μπορεί να επιλέξει να πάρει αυτή την άδεια ή να την χάσει αν δεν την πάρει και πιστεύω πως αυτό έχει επιτυχία και θα επηρεάσει θετικά και αλλού τομεί, όπως και παράδειγμα την αγορά εργασίας. Έτσι θα, θα αναγκάσουν τους πατέρες να συμμετέχουν πιο ενεργά στις ζωές των παιδιών τους. Βέβαια, σχετικά με τις ε, μισθολογικές και συνταξιοδοτικές ε, ε, διαφορές, ε, σίγουρα υπάρχουν οι γυναίκες έχουν το 60% των συνταξιοδοτικών απολαβών των ανδρών. Χρειάζεται λοιπόν να αλλάξει αυτό. Και επίσης χρειάζεται να γίνει ένα σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην εργασία επιπληρωμή και στην άμεση εργασία. Αυτά προς το παρόν. Ελπίζω να κατάφερα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και θα χαρώ πολύ να συνεχίσω την συνεργασία με όλους εσάς που επιθυμείτε μια ισχυρότερη δέσμευση για την ισότητα των φίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ευχαριστώ Υπουργέ. Εύχομαι να σας ξαναβούμε σύντομα. Allora, riprendiamo la nostra riunione, affrontiamo adesso il punto 5, eh, presentiamo due studi. Περνάμε στο σημείο 5, έχουμε δύο μελέτες. Η μία έχει προετοιμαστεί από την ε, Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων 3 ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, εμπειρικές συλλογές πληροφοριών σχετικά με την έκθεση η οποία προετοιμάζεται ε, στις 15 Οκτωβρίου να κατατεθεί ε, στην ε, Επιτροπή μας έκθεση πρωτοβουλίας εξωτερικοί παράγοντες στην γυναικεία επιχειρηματικότητα. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα ακούσουμε την εμπειρική βάση θα έλεγα τα στοιχεία τα επιμέρους τα οποία θα χρησιμεύσουν στην εισηγήτρια να συγγράψει τη σημαντική έκθεσή της, μια έκθεση που για πρώτη φορά προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα θέματα που έχουν οι γυναίκες στην Ευρώπη, ε, αντιμετωπίζουν τεράστια εμπόδια. Θα δώσω λοιπόν στην κυρία Μακράκεν το λόγο, η οποία είναι συνεργάτης της Opchit Research, ζητήθηκε η μελέτη αυτή από την δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Η κυρία Μακράκιαν είναι διευθύντρια στο τμήμα έρευνας της Omchit Research και έχει κάνει πολλές εμπειρικές μελέτες για το Ηνωμένο Βασίλειο, για αρκετές ΜΚΟ και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Είναι ευτυχιούχος του lc e. ε, the micro. Yeah, yes, that'd be good. Thank you very much. Okay, thank you for the introduction and for the invitation. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Κοιτάξαμε τα ποσοστά της γυναικείας επιχειρηματικότητας ε, στην Ευρώπη, όχι γενικότερα, αλλά ειδικότερα την φύση της επιχειρηματικότητας και τις διαφορές της γυναικείας επιχειρηματικότητας, τις ε, διαφορές τα ποσοστά μεταξύ ανδρικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας και το ε, είδος των επιχειρήσεων που δημιουργούν οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω με συντομία το θέμα μας λοιπόν. Αυτή η διαφάνεια μας δείχνει τα γενικότερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης. Τα ποσοστά αυτά χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματικότητα. Δεν είναι πανάκια βέβαια αυτά τα στατιστικά στοιχεία, όμως σας δίνουν μια γενικότερη εικόνα του τι συμβαίνει με την αυτοαπασχόληση, ε, τουλάχιστον μέχρι το 2014. Τα ποσοστά των 24 ε, χωρών λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπου αυτά. Αν δούμε όμως προσεκτικά τα ποσοστά αυτά θα δούμε πως υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες στις 24 αυτές χώρες. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ε, επιχειρήσει ανδρών και γυναικών. Βλέπουμε ότι οι άνδρε έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό αυτοαπασχόληση από τι γυναίκε. και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ε, στα ποσοστά ανδρών και στα ποσοστά γυναικών. Μπορούμε λοιπόν, σε... συνοψίζοντας, να πούμε ότι περίπου το 14% των εργαζόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτοαπασχολούμενοι. Στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη υπάρχουν μεγαλύτερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης. Βέβαια δεν συμπεριλαμβάνουμε τις περιοχές που έχουν υψηλά ποσοστά γεωργίας και άτυπης εργασίας. Στη Βόρεια Ευρώπη τα ποσοστά αυτοπασχόλησης είναι μικρότερα. Όμως, αν κοιτάξουμε ακόμα πιο προσεκτικά και δούμε τις ε, διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα και την επιχειρηματικότητα, θα δούμε ότι μόνο το 1 τρίτο περίπου το, των 40 εκατομμυρίων ε, αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών δηλαδή, είναι γυναίκε, τουλάχιστον το 2012. Επίση, βλέπουμε ότι τα ποσοστά αυτοαπασχόληση για τις γυναίκες ε, βρίσκονται πολύ πίσω από τα αντίστοιχα των ανδρών σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και υπάρχουν κάποιε διαφορέ. Οι μεγαλύτερε διαφορέ παρατηρούνται στην Ιρλανδία, τη Σουηδία και τη Δανία. Επίση, όμω και στην ε, Σλοβακία οι, με, οι μικρότερες ε, διαφορές είναι στο Λουξεμβούργο και ίσως στην Πορτογαλία. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη διαφοροποίηση σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Επίσης, Υπάρχουν διαφορές στην ερμηνεία του τι, είναι, του τι καθιστά κάποιον επιχειρηματία. Αν δούμε τις χώρες του ΩΣΑ θα παρατηρήσουμε ότι οι γυναίκες είναι ιδιοκτήτριες περίπου του 1 τρίτου των ε, επιχειρήσεων στις πόλεις. Όμως, κοιτάζοντας ε, λίγο προσεκτικά την κοινωνική επιχειρηματικότητα, Δηλαδή όχι την κερδοσκοπική απασχόληση αλλά την μη κερδοσκοπική, την κοινοφελή απασχόληση θα δούμε ότι υπάρχουν περισσότερη ε, ομοιομορφία. Υπάρχουν βέβαια διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις, ε, στα κρατημέλη, όμως φαίνεται ότι οι γυναίκες με υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης ε, έχουν ίδια ποσοστά αυτοαπασχόλησης και επιχειρηματικότητας με τους άντρες. Η διαφορά μεγαλώνει ε, όσο χαμηλώνει το μορφωτικό επίπεδο. Αυτό για μας σημαίνει μια μεγάλη απώλεια για την οικονομία. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου μορφωμένες γυναίκες δεν ε, δημιουργούν επιχειρήσεις. Επίσης, οι υπηρεσίε που παρέχουν οι γυναίκε στην κοινωνία είναι πάρα πολύ υψηλέ. Οι γυναίκε που ιδρύουν κοινοφελεί επιχειρήσει είναι περισσότερο πιθανό να δημιουργήσουν και κάποια ε, κερδοσκοπική επιχείρηση. Για, πολλούς, ε, λοιπόν, ε, για πολλές γυναίκες το να ε, δημιουργήσουν μια κοινοφελή μη κερδοσκοπική επιχείρηση είναι κάπως σαν βάπτισμα του πυρός για να κάνουν τη δική τους επιχείρηση αργότερα. Μετά, σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και το φύλλο, βλέπετε εδώ αυτή τη διαφάνεια που ε, αναφέρει τα χαρακτηριστικά των ε, γυναικείων επιχειρήσεων. Βλέπουμε πως οι γυναίκες τείνουν να είναι επικεφαλής μικρότερων επιχειρήσεων με μικρότερο τζίρο και ε, μικρότερες ε, πιθανότητες ανάπτυξης. Επίσης, οι τομεί στους οποίους δραστηριοποιούνται γυναίκες και αρχίζουν και δημιουργούν κάποια επιχείρηση θεωρούνται από τις τράπεζες, από πολλές τράπεζες τουλάχιστον, ως λιγότερο κερδοφόρες, με λιγότερο δυναμικό ανάπτυξης. Επίσης, βλέπουμε πόσο πολλές γυναικείες επιχειρήσεις βασίζουν, έχουν έδρα το σπίτι των γυναικών αυτών Είναι δηλαδή επιχείρηση του ενός ε, απασχολούμενου και βλέπουμε πως οι επιχειρήσεις αυτές ε, διαστηριοποιούνται σε τομείς που έχουν ε, χαμηλότερη προστιθέμενη αξία. Βλέπουμε πως περίπου 5 έως 15% των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας έχουν δημιουργηθεί από γυναίκες και αυτά το έβριμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, στα δεξιά της διαφάνειας αυτής βλέπουμε ότι οι γυναίκες όταν οι ίδιες μιλούν για τις ε, επιχειρήσεις τους έχουν χαμηλότερες προσδοκίες ε, από αυτές. Ε, προσδοκίες για χαμηλότερο τζίρο δεν πιστεύουν ότι θα εξελιχθούν, ότι θα αναπτυχθούν, θα μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις τους. Επίσης έχουν και μικρότερες φιλοδοξίες σε σχέση με τους άντρες για να μεγαλώσει η επιχείρησή τους. Αυτό βασίζεται σε διάφορα στατιστικά δεδομένα που αποκομίσαμε μετά από έρευνες. Επίσης, όταν ζητήθηκε από τις γυναίκες να αξιολογήσουν το επίπεδο καινοτομίας της επιχείρησής τους, ε, αυτές το αξιολόγησαν όσο χαμηλότερο σε σχέση με τους άντρες. Τώρα, ας δούμε τα αποτελέσματα ε, της έρευνάς μας σχετικά με την σχετική νομοθεσία. Νομοθεσία η οποία θα επηρεάσει τα ποσοστά της ανδρικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας. Ε, τα σημαντικότερα βρήματα βρίσκονται σε αυτήν την διαφάνεια. Υπάρχουν προσπάθειες να ε, αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα όσον αφορά τι άδειε μητρότητα ή αυτοαπασχολούμενε γυναίκε. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, για παράδειγμα η αυτοαπασχολουμενε γυναικε εχουν γινει σημαντικα βηματα σχετικά με την αυτοαπασχόληση, η οποία πρεσβεύει η συμμεταχείριση ανδρών και γυναικών και η συμπρόσβαση στις υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και τις ε, τραπεζικές υπηρεσίε. Υπήρξαν επίσης κάποιες ε, θετικές εξελίξεις που προώθησαν την ισότητα, για παράδειγμα ε, οδηγίες οι οποίες προώθησαν ε, μέτρα υπέρ της ισότητας. Τώρα, απαγορεύονται φυσικά οι διακρίσεις ανάλογα με το φύλλο. Όμως, σε μία έρευνα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουμε την άμεση, ε, τις άμεσες από τις σε διακρίσεις. Υπάρχει ένα ψήφισμα του 2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου παρατηρείται ε, δυστυχώς η ανισότητα στην ε, πρόσβαση των γυναικών στη χρηματοδότηση, ιδιαίτερα των γυναικών που είναι μονογονεϊκές οικογένειες. Όσον αφορά τώρα την επιτυχία των γυναικείων επιχειρήσεων. Είχαμε κάποιες μελέτες από την Τσεχία όπου διεξήγαμε διάφορες ε, έρευνες. Είδαμε ότι υπάρχει κάποιος ε, δισταγμό σχετικά με την χρηματοδότηση των γυναικείων επιχειρήσεων. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά κάποια βασικά παραδείγματα. Τσεχία. Οι γυναίκες επιχειρηματίες Κάτι που είδαμε σε πολλές απαντήσεις, ζητούν χρηματοδότηση σπανιότερα από ότι οι άνδρες και όταν το κάνουν αυτό ζητούν χαμηλότερα δάνεια. Αυτό ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι οι ίδιες οι γυναίκε δεν θέλουν να ζητήσουν πολλά χρήματα, δεν θέλουν να ε, αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο και αυτό συνήθως αποθεί τους δανειστές διότι όταν δανείζουν μικρότερα ποσά έχουν και μικρότερα κέρδη. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε ότι μια γυναίκα επιχειρηματίας μας, είπε ότι την θεωρούσαν ενόχληση οι τράπεζες, θεωρούσαν ότι δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν με την περίπτωσή της. Τώρα, σχετικά με τις άδειες μητρότητας, γονικές άδειες, εδώ παρατηρήσαμε ότι όταν μια γυναίκα κάνει αίτηση για δάνειο στην τράπεζα, υφίσταται διακρίσεις σχετικά ε, με, τη γονική άδεια. Τώρα, επίσης, υπάρχει και μία αναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, ε, δηλαδή η συλλογική, συμμετοχική χρηματοδότηση, το crowdfunding, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μία αναλλακτική λύση για να ε, βρεθεί κεφάλαιο. Υπάρχουν επιπρόσθετες προκλήσεις για τις γυναίκες επιχειρηματίες για παράδειγμα το ότι είναι δυσανάλογο το βάρος ε, που έχουν για την ε, φροντίδα των παιδιών. Επίσης υπάρχουν διαφορές στα επίπεδα αισιοδοξία που τις εμποδίζουν από το να έχουν μια επιτυχημένη επιχειρηματική σταδιοδρομία. Τώρα, άλλη ε, περίπτωση Ιταλία οι γυναίκες τείνουν να δημιουργούν επιχειρήσεις σε παραδοσιακά γυναικοκρατούμενους τομεί, όπως για παράδειγμα αισθητική, υπηρεσίες καθαρισμού, υπηρεσίες ε, υγείας. Αυτοί όμως ε, οι τομέί είναι λιγότερο ελκυστικοί για τους ε, χορηγούς, για τους χρηματοδότες. Βέβαια, οι γυναίκε δραστηριοποιούνται εκεί επειδή έχουν συνήθω μεγαλύτερη εμπειρία. Τώρα, ε, τα, μέσο, το μέσο δάνειο στους, ε, στις ε, γυναίκες επιχειρηματίες είναι κατά πολύ χαμηλότερο από το μέσο δάνειο που παίρνει ένας άνδρας επιχειρηματίας. Κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θεώρησαν γυναίκες επιχειρηματίες ως πάρα πολύ σημαντικά για να πετύχουν ήταν καταρχάς η πρόκληση που αποτελεί το να φτιάξεις τη δική σου επιχείρηση. Αυτό εκπλήρωση που σου δίνει η δημιουργία μιας επιχείρησης. Και στην περίπτωση της Ιταλίας η οικογένεια στήριξε και συναισθηματικά και ε, οικονομικά τις ε, γυναίκες επιχειρηματίες και οικονομικά λοιπόν αλλά και ε, με την φροντίδα παιδιών, με την ανάληψη διάφορων φορτίων που είχα, έχουν επομιστεί οι γυναίκες. Τώρα υπάρχει η περίπτωση της Σουηδίας. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν και τα venture capital από τις κεφαλαιαγορές και όχι μόνο τράπεζες. Οι επενδυτές μετά από αυτά τα οποία είπα, οι οποίοι είναι άνδρες συνήθως, ή αυτοί που αποφάζουν, αποφασίζουν συγγνώμη, για το πού θα δοθούν οι επενδύσεις, έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους άνδρες συνομιλητές. Και υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές ε, ε, στα δίκτυα τα επιχειρηματικά ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Γενικά τα δίκτυα τα οποία ελέγχονται από γυναίκες έχουν μικρότερη επιρροή και οι γυναίκες έχουν ε, λιγότερες γνωριμίες συνήθως από ότι οι άνδρες έτσι ώστε να μπορέσουν να συναντηθούν με venture capitalists που είναι απαραίτητοι για την χρηματοδότησή τους. και γενικά ενδιάμεσα στελέχη έδειξαν ότι υπάρχει ένας δι... Ένα δισταγμός από πλευράς των γυναικών που λειτουργούν συντηρητικά και δεν θέλουν να δημιουργηθούν κίνδυνοι οικονομικοί για αυτούς και την οικογένειά τους. Ε, για την χρηματοδότηση του χρέους στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει πιο σοβαρό πρόβλημα. Ε, δεν αναζητούν χρηματοδότηση για κάλυψη χρέους και όταν το κάνουν ζητούν λιγότερα χρήματα. κάτι το οποίο βλάπτει τη δυναμική της επιχείρησής τους. Με τα venture capitals γενικά οι γυναίκες έχουν μικρότερες εμπειρίες, λιγότερες εμπειρίες και ως εκ τούτου μικρότερη έκθεση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες υπάρχει ισχυρή κοινωνική επιχειρηματικότητα Παρ' όλα αυτά ο τομέας αυτός ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σχετικά περιορισμένος. Οι γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο διστάζουν να πούν για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν λόγω του ότι είναι γυναίκες προσπαθούν από μόνες τους να ξεπεράσουν τα εμπόδια αυτά και θεωρείται κατόρθωμα όταν το πετυχαίνουν. Πρέπει να είναι εξαιρετικές γυναίκες για να μπορέσουν να πετύχουν στον επιχειρηματικό κόσμο ενώ ένας μεσαίος άνδρας ε, είναι στην ίδια κατάσταση υποτίθεται με αυτές. Υπάρχουν πολλές επιμέρους μελέτες που δείχνουν ότι υπάρχουν ε, και στις αμοιβέ των επιχειρηματιών διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες εις βάρος των γυναικών. Πάντως το βασικό πρόβλημα είναι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Οι γυναίκες όπως είπα δεν αναζητούν χρηματοδότηση τόσο συχνά όσο οι άνδρες και τόσο πολύ όσο οι άνδρες αλλά υπάρχει μια κάποια σχέση ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά στον τομέα της χρηματοδότησης. Γυναίκες θεωρούν ότι δεν είναι για αυτές οι χρηματοδοτικές δυνατότητες και γι' αυτό δεν τις αναζητούν. Υπάρχουν επίσης και σημαντικά διαφορετικά θέματα που παρεμποδίζουν την πρόσβαση των γυναικών στην χρηματοδότηση. Είπαμε ότι και σε επίπεδο κάλυψης χρέους και σε επίπεδο venture capital οι γυναίκες έχουν μικρότερη εμπλοκή. Αυτό αντικατοπτρίζει έτσι και αλλιώ τις διακρίσεις ε, τις οποίες υφίστανται οι γυναίκες γενικά και στην ίδια την αγορά εργασίας. Γενικά έχουν μικρότερη εξουσία, και ε, οι οικογενειακές επίσης φροντίδες είναι ένα επιπλέον εμπόδιο για τις γυναίκες επιχειρηματίες. Αυτό αποδεικνύεται, αποδείχθηκε στη μελέτη με πολλούς τρόπους, ποιοτικούς τρόπους που είναι δύσκολο να επιδειχθούν. Αλλά πάντως για τις γυναίκες υπάρχουν λιγότερο ευνοϊκοί όροι και αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο στις επιχειρηματικές συναντήσεις. Οι συστάσεις μας λοιπόν σε σχέση με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ότι απαιτούνται νέα προγράμματα έτσι ώστε οι τράπεζες να δανείζουν σε εταιρείε που ανήκουν σε γυναίκες και σε επίπεδο μικροχρηματοδότησης και σε επίπεδο εγγύησης δανειοδότησης. Ιδιαίτερα σε τομείς όπου υπάρχει αργή επιστροφή και απόσβεση, σε τομείς όπου ε, κυριαρχούν οι άνδρες υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα διαφορετικά και κάποιες διακρίσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι γυναίκες να υπάρξει βοήθεια για τη διεύρυνση των γυναικείων επιχειρηματικών δικτύων. Μια επιχειρηματία στη Σουηδία σαν παράδειγμα συναντήθηκε με πάρα πολλούς άνδρες και γυναίκες για να γνωριστεί και να συζητήσει μαζί τους έτσι ώστε να μπορέσει να αποσύρει κάποια από τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Και απαιτείται περαιτέρω έρευνα έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανόηση και των μέτρων έμεσης διάκρισης της βάρος των γυναικών επιχειρηματιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μακκράκεν. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μόσκα υπεύθυνο για θέματα φύλων στο Ινστιτούτο AG που είναι το υπεύθυνο για την ισότητα των πολιτών. Ο κύριος Μόσκα εργάζεται στο Ινστιτούτο αυτό από το 2011, είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των εργασιών του Ινστιτούτου αυτού για τη διάδοση των χρηστών πρακτικών. Έχετε το λόγο κύριε Μόσκα. Καλησπέρα σε όλου. Ευχαριστώ εσάς και την Επιτροπή σα που με προσκαλέσατε εδώ για να παρουσιάσω τι εργασίε του Age. Ευχαριστώ την Έρικα που με ενέπλεξε. Ελπίζω να είναι η πρώτη από μια σειρά από περαιτέρω επαφές. Ευχαριστώ και την επιμελητία και θα περάσω τώρα στην αγγλική γλώσσα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, να διαβάζει κανείς τα πορίσματα αυτής της έκθεσης. Νομίζω ότι είναι συμπληρωματική η δουλειά που κάνουμε. Θα ήθελα σύντομα να σας ενημερώσω για το τι κάνουμε εμείς ε, στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Ε, ε, πονήσαμε αυτή την έκθεση στα πλαίσια της εργασίας ε, της ΕΓΚΕ με την ελληνική προεδρία. Εφτά μήνες διήρκησε και συλλέξαμε στοιχεία σε σχέση με τη σύσταση επιχειρήσεων το 2011 και αυτή είναι ακριβώς μία από τις μαλαμβανόμενες εκθέσεις που ε, τη ΣΥΟΣ. Θα ήθελα εν συντομία να σας την παρουσιάσω. Σας έχω ήδη στείλει ε, τους πόρους και είναι πραγματικά στη διάθεσή σας αν λείπει κάτι. Εγώ θα ήθελα ε, σε τρία σημεία να επικεντρωθούμε που είναι και τα βασικά επιτεύγματά μας μέσα από αυτή την έκθεση. Δηλαδή ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κατά τη διάρκεια αυτές τις διαδικασίες και να ε, συνάψω και κάποια συμπεράσματα ούτως ώστε ενδεχομένω να καταλήξουμε και συστάσεις για την προώθηση ε, της συμμετοχής των γυναικών, της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας αλλά και την προώθηση της γυναικής επιχειρηματικότητας. Ποια είναι τα βασικότερα επιτεύγματα. Ολοκληρώθηκε το Μάιο 2014 η έκθεση, σχεδόν έχει περάσει ένας χρόνος δηλαδή. Και βάσει του στόχου μας ε, θέλουμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη ιδίων ιδενοτήτων, capacity building, αλλά και την ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων για τα θέματα αυτά, ούτως ώστε να τονωθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, κυρίως ως προς την γυναική επιχειρηματικότητα. Ήταν αρκετά εντατική αυτή η δουλειά μπορώ να πω. Η παρουσίαση δε των αποτελεσμάτων και διάδοσή τους ε, ήταν ευρύτατη. Δεν θα ήθελα τώρα να παριθμίσω όλες τις προσκλήσεις που λάβαμε για να παρουσιάσουμε τα ε, αποτελέσματα. Να σας πω μόνο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει και πλατφόρμα για την ανταλλαγή βαλτίστων πρακτικών φυσικά μας κάλεσε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα και το ίδιο και εμπλεκόμενοι φορείς ε, που ασχολούνται στον τομέα κατάρτισης πολιτικής, το West Network από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ επιχειρήσεων κάνει επίσης σε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά και ε, με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς ε, είμαστε σε διαρκή επαφή για την ανταλλαγή και τη διάδοση βελτίστων προκτικών ε, και έχουμε και σε εθνικό επίπεδο δράση των εθνικών κυβερνήσεων μέσα από σημεία επαφής, στρατηγική για την πρόθεση της γυναικής επιχειρηματικότητας, Λιθουανία, στη Ρήγα συγκεκριμένα έγινε διάσκεψη για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών, Ιταλία, Εθνική Βάση Δεδομένων για τα θέματα ισότητας των δύο φύλων και στην Ισπανία σε αρχές του 2015 ε, το ε, Εθνικό Ινστιτούτο διοργάνωσε και την ε, Εθνική μέρα για τη γυναική επιχειρηματικότητα. Βασιζόμαστε σε αυτά που μαθαίνουμε και αυτό που ε, διαθέτουμε είναι από συγκεκριμένες αυτές λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν ε, σε κράτη-μέλη. Επίσης, μία απλή αλλά και πάρα πολύ εύστοχη μεθοδολογία για τον εντοπισμό των βελτίστων πρακτικών. Αυτό είναι ένα άλλο επίτευγμά μας. Δεν θεωρούμε, ε, δεν ισχυριζόμαστε ότι μπορούμε να χαρτογραφήσουμε όλες τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη ή ότι έχουμε εντοπίσει όλες ε, τις ε, καλές πρακτικές. Όμως έχουμε ολοκληρώσει τη διαβούλευση με ευρύτατο το δίκτυο εμπλεκομένων φορέων για να εκπονήσουμε την έκθεση και σίγουρα υπάρχει αξιακή αξία. Μπορούμε να αντιλησουμε διδάγματα από αυτή την έκθεση, να δούμε ποια είναι τα εφιστάμενα προβλήματα, τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να δούμε τι ε, τελικά αποτελεσματικό, τι οδήγησε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η μικρή μας συμβολή στη συζήτηση λοιπόν θα σχετιστεί περισσότερο με τις βέλτιστες πρακτικές που προέρχονται από 10 κράτη-μέλη και τρία συγκεκριμένα ε, εργαλεία, το networking, η δικτύωση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η πρόσβαση στα κονδύλια, χρηματοδότηση δηλαδή. δύσκολο μετά από όλες αυτές τις παρεμβάσεις ε, να κάνω μια παρουσίαση που θα μπορέσετε να σχετίσετε στο μυαλό σας με όσα έχουν υποθεί. Θα προσπαθήσω όμως ε, να ακολουθήσω ε, το μύτο των προηγούμενων παρουσιάσεων. Τι προκύπτει λοιπόν από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με τα δίκτυα των εμπλεκομένων φορέων και των οργανώσεων. Ποια είναι τα κολλήματα που ακόμη φύστανται. Ήσασταν ξεκάθαροι εσείς στην παρουσίασή σας για αυτό το ευρύ φάσμα εμποδίων που είναι μια πραγματική τροχοπέδη για τις γυναίκες κατά της οικονομικής και κοινωνικής χειραφέτησης και της πρόσβασής στην αγορά εργασίας αλλά και στην επιχειρηματικότητα. Τέσσερα είναι τα βασικά στοιχεία για μας. Πρώτον πρέπει να γίνει χαρτογράφηση των βιωμάτων. Δεύτερον, Το θέμα των πόρων ξέρουμε ότι ε, σε κάποια δίκτυα, σε κάποιες χώρες αυτό ήδη συμβαίνει. Αλλά ακόμα θα ήταν όπως είπε και η Σουηδή Υπουργός ε, είναι να έχουμε μια γενικότερη κατεύθυνση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ώστε όλα τα κράτη-μέλη, όλε τι περιφέρειες να ε, συμβάλλουν σε μια κοινή προσπάθεια. Η ανταλλαγή λοιπόν βελτίστων πρακτικών, η συλλογή ε, δεδομένων, η έρευνα είναι ε, στοιχεία σημαντικά για να ε, κατανοήσουμε τις πρακτικές, φυστάμενες πρακτικές σε σχέση με τη γυναική αποχειρηματικότητα. Συστηματική λοιπόν συλλογή στατιστικών δεδομένων, δεδομένων που έχουν αποδομηθεί κατά κάποιο τρόπο αφαιρώντας την διάσταση των δύο φύλων. Μόνο έτσι μπορούμε να καταπολεμήσουμε το μισθολογικό χάσμα που συνήθως είναι εις βάρος των γυναικών. Η παρακολούθηση και η αποτίμηση είναι εξίσου σημαντικές για να κατανοήσουμε ποιος ήταν ο αντίκτυπος των πολιτικών, ποια είναι η επιστροφή, αν θέλετε, της επένδυσης ε, που έχουμε κάνει μέσω των πολιτικών επιτόπου. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Ιδίως μεσού τη κρίση. Ας μην μιλήσουμε για το κόστος των διοχετεύουμε κονδυλά, μιλήσουμε για επένδυση, διότι εκεί που έχει γίνει η ανάλυση, η αξιολόγηση, παρακολούθηση, η αποτίμηση, είναι έχει προκύψει με σαφήνεια ότι αυτή η επένδυση είναι υποφελής για ολόκληρη την κοινωνία και για τα δύο φύλλα για μας. Αυτό θα πρέπει να είναι ε, ένα χειρό και εναργές μήνυμα, ούτως ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη τελικά υποστήριξη για την πολιτική ε, πρόθεση ισότητας των δύο φύλων. Τώρα η βιωσιμότητα ας συνειδητοποιήσουμε ότι πέρα από τα αρχικά κονδύλια για τη σύσταση μιας επιχείρησης, ε, όπως μας είπατε και εσείς, ε, υπάρχουν πολλά περαιτέρω βήματα. Αυτό είναι το πρώτο λιθαράκι, αν θέλετε, το πρώτο βήμα. Χρειαζόμαστε υπηρεσίες υποστήριξης πέρα από την υποδομή, χρειάζεται υποστήριξη για τη δικτύωση, για την ανάπτυξη των προσωπικών, διαπροσωπικών δεξιοτήτων, των περίφημων soft skills, ούτως ώστε να ευρεωθούν οι νέες επιχειρήσεις, ε, να σταθεροποιηθούν. Για την ανεργία των ε, γυναικών ε, έχουμε κάνει μελέτες στον επιχειρηματικό κόσμο. Δεν θα μπω σε συγκεκριμένα παραδείγματα, όμως μπορώ να σας μιλήσω για μια γυναίκα που έκανε που είχε ένα ιδιαίτερο όραμα για τις συνεταιρικές αυτές τράπεζες στην Κύπρο Αυτό το παράδειγμα μας δείχνει ότι ε, κάνοντας αυτή την επένδυση έχουμε ανάπτυξη ε, που είναι υποφελής ε, και για τα δύο φύλλα και για το σύνολο της κοινωνίας. Πρέπει να αποτινάξουμε αυτό, αυτή την ιδεολογική φόρτιση και να θεωρηθεί αυτονόητο πως χρειάζεται η ανδρική συμβολή στην προσπάθεια. Νομίζω ότι εξήγησα και τα πέντε μου λεπτά. Ε, ας καλύτερα σταματήσω για να υπάρχουν και, αφού πρώτα αντλήσω κάποια συμπεράσματα, για να ε, έχουμε και χρόνο για τις ερωτήσεις. Συμπεράσματα λοιπόν. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια νούμερα. Μετά από τη διαδικασία διαβούλευσης, με τους εμπλεκόμενους, τους ενδιαφερόμενους φορείς των εθνικών φορέων αλλά και δίκτυα επιχειρηματιών, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, ένα ευρύ φάσμα ε, φορέων, νομίζω, καταλήξαμε όλοι σε κοινά συμπεράσματα. Ποια είναι αυτά, πρώτον. Τι να πω τώρα, θα επανεφεύρω τον τροχό, αλλά τέλος πάντων ε, είναι σημαντικό να πω πως όταν μιλάμε για την ε, γυναική επιχειρηματικότητα θα πρέπει να βλέπουμε ένα να έχουμε μια ευρέτερη εικόνα μπροστά μας. Πέρα από τις γυναίκες υπάρχουν διαφορετικές προσδοκίες, διαφορετικά ταλέντα, διαφορετικές δεξιότητες, διαφορετικά συμφραζόμενα, διαφορετικά στοιχεία και όλες οι διαστάσεις κάθε συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να συνυπολογίζονται για να καλύψουμε τις ανάγκες. Ε, δεύτερον, ο στρατηγικός ρόλος που έχουν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όχι για να ε, ευλογήσουμε τα ε, μουσια μας αλλά είναι απαραίτητο για να επιτύχουμε, να υλοποιήσουμε αυτούς τους οικονομικοκοινωνικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι άλλο που έχει αναγνωριστεί ως ε, κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης ε, είναι η δεκτήωση και οι πρακτικές mentoring, ε, ώστε να υπάρξει μια πλαισίωση, μια υποστήριξη μέσω ε, μιας ε, πλατφόρμας ώστε να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση ε, των νέων επιχειρηματιών. Ο Υπουργό αναφέρθηκε στη σύμβαση του 95 του Πεκίνου, στη δήλωση του Πεκίνου μάλλον του 95 και μας μίλησε για το mainstreaming, ένας από τους βασικούς πυλώνες και παραμένει αυτό ένα Κύριε σημασία εργαλείο για να καλύψουμε τις ανισότητες που εξακολουθούν να παρατηρούνται. Μιλήσαμε για το ρόλο των, των ε, γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των ε, εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρεών Αλλά για την κάλυψη αυτού του χάσματος είναι, παραμένει, ήταν και παραμένει θεμελιώδης ο ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι άλλο που ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον στην ανάλυση που κάναμε ήταν ε, η προσέγγιση που σχετίζεται με την κινητοποίηση όχι μόνο των παραδοσιακών ε, φορέων, τα ΜΜΕ, τραπεζικό τομέα των οργανώσεων, όχι, αλλά ε, το φεμινιστικό κίνημα κινητο, διαφορετική αλλά μέσα κινητοποίηση ε, της κοινότητας και συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει άλλος τρόπος να αντιληφθούμε τις συγκεκριμένες ανάγκες ε, που υπάρχουν αλλά και να ε, επιτύχουμε την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση για να καταλύσουμε τους φραγμούς που ακόμη υπάρχουν. Αναφερθήκατε εσείς ε, στα, στα στερεότυπα. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν προκαταλήψεις, όχι μόνο στερεότυπα, για την ε, χρηματοδότηση των ε, γυναικείων επιχειρηματικών σχεδίων. Έτσι μπορούμε να άρουμε κάποιους από αυτούς τους φραγμούς, λοιπόν. Με εναλλακτικά μέσα ε, κινητοποίησης. Α, ναι, και ο υπουργό μας μίλησε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις συμβουλές για την επαγγελματική σταδιοδρομία. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθούν οι μονομένες φιλοδοξίες των νέων επιχειρηματιών μέσω από υπηρεσίες υποστήριξης ε, και ε, ενίσχυση επίσης των ταλέντων μέσα από την αύξηση της αποσχολησιμότητας. Ε, πέρα από αυτά τα στερεότυπα, πέρα από αυτά τα από αυτές τις αποφάσεις που ήδη έχουν αποτύχει πολλά και στην αγορά εργασίας και έχουν οδηγήσει στην σημερινή απόγνωση για την επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση από πρόωρα στάδια για την ε, δημιούργηση των ε, δεξιοτήτων, για την οικοδόμηση αυτής της ε, επιχειρηματικής νοοτροπίας νομίζω ότι αυτό μας το δείχνουν και άλλες εκθέσεις, η επιχειρηματική νοοτροπία όχι μόνο επιτρέπει στις γυναίκες ε, να κάνουν το βήμα και να συστήσουν την επιχείρηση αλλά και αντιμετωπίζουν δύο βασικές προκλήσεις, την φτώχεια. Ε, μίλησε η υπουργό ε, για την... για το πρόβλημα του μυθολογικού χάσματος, δηλαδή αυτό είναι θα μεγαλύτερο ακόμη άχθος για το ασφαλιστικό σύστημα και παγιοποιείται η φτώχεια πρώτον και δεύτερον για, ακόμη και για τη βία κατά των γυναικών ε, μας βοηθά η οικοδόμηση του επιχειρηματικού πνεύματος για την αυξημένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας ε, με μία θέση εργασία είναι σε καλύτερη θέση η γυναίκα οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει την απειλή τη σεξουαλική βία. Δεν θέλω να μπω ε, σε συγκεκριμένα παραδείγματα, με τα χαρά σε να σα δώσουμε όλα τα στοιχεία για τη δουλειά και την εμπειρία που έχουμε, όχι μόνο σε αυτόν τον τομέα αλλά και σε όλου. Θα ήθελα να τονίσω ότι είμαι στη διάθεσή σας ε, αν ενδιαφέρεστε για αυτά τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μόσκα. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο εμπειρογνώμονες γιατί μας έδωσαν τη δυνατότητα να αρχίσουμε ε, την ε, συζήτηση πάνω στην προετοιμασία αυτής της έκθεσης η οποία πραγματικά θα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι πραγματικά πολύ επίκαιρο και σημαντικό ζήτημα. Είμαι η εγώ προσωπικά και ως εισηγήτρια πρέπει να πω ότι μας είπατε πάρα πολύ σημαντικά ε, πράγματα. Καλύψατε πολλά θέματα, εξάλλου είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο και πολύ σχηδές. Επίσης, Θα ήθελα να σας πω πως ε, λυπάμαι για το ότι δεν είχαμε μεγάλη προσέλευση σήμερα. Είχαν αρκετή προβλήματα με τις πτήσεις τους και δεν κατάφεραν να έρθουν. Όμως ε, στις 15 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει αυτή η Επιτροπή ξανά και να είστε σίγουρος ότι μας δώσατε πολύ τροφή για σκέψη. Θέλουμε όλοι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δηλαδή υπαρκτές απτές λύσεις για τη βελτίωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και τους δύο πάρα πολύ. Μας δώσατε πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Χρησιμοποιήσατε μια ιδιαίτερα χρησιμοποιητική προσέγγιση έτσι ώστε τα στοιχεία που μας δώσατε να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερα. Είναι πραγματικά ε, εκπληκτικά αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή για το 2000 12 που μας είπατε ότι μόνο το 29% των ε, ε, αυτοαπασχολούμενων είναι γυναίκες. Πιστεύω πως σήμερα υπάρχει κάποια βελτίωση, εξακολουθεί όμως να υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά γυναικείας και επιχειρηματικότητας. Όμως με βάση τα στοιχεία που μας δώσατε μπορούμε να σχεδιάσουμε για το μέλλον και να εστιάσουμε στις ε, περιπτώσεις όπου εσείς ε, αναφερθήκατε. Μας είπατε ότι οι γυναίκες επιλέγουν συγκεκριμένους ε, τομείς αυτοαπασχόλησης με χαμηλότερο τζίρο, χαμηλότερο εισόδημα, ενώ οι άντρες συνήθως επιλέγουν τους τομείς των υποδομών, της πληροφορικής, της υψηλής τεχνολογίας. Αυτό λοιπόν μα έδωσε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα αξιοποιήσει αυτά και χρειάζεται φυσικά να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών στη χρηματοδότηση. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή μας, πρέπει όμως να δώσουμε απαντήσεις. Πώς να βελτιωθεί η πρόσβαση, πώς να διερευνήσουμε εναλλακτικού τρόπους χρηματοδότησης, για παράδειγμα την ε, μικροχρηματοδότηση που είναι πολύ σημαντική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι πρέπει να αλλάξουν οι πρακτικές έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Και η υπουργό ε, της ε, Σουηδίας που ήταν πριν από λίγη ώρα εδώ μας έδωσε το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό. Η Σουηδία είναι πολύ πιο μπροστά από τις άλλες χώρες. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλοί φραγμοί που πρέπει να ξεπεραστούν ακόμα για να επιτευχθεί η πραγματική ισότητα των φύλων. Υπάρχει ένα στίγμα αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, στην γυναικεία επιχειρηματικότητα. Υπάρχει Υπουργείο αρμόδιο για τις ίσες ευκαιρίες, όμως αυτό δείχνει ότι πρέπει να γίνουν ακόμα πάρα πολλά για την ισότητα. Και σίγουρα δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στα λόγια. Χρειάζεται νομοθεσία που θα εφαρμόζεται. Χρειάζεται αυτό να, αυτές οι προσπάθειες να φαίνονται και στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και αυτά σας ε, τα λέω και ως ε, Ευρωβουλευτής και ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν ξανά να σας ευχαριστήσω για όσα μας ε, παρουσιάσατε και θα ήθελα επίσης να σας συζητήσω συγγνώμη για τους συνάδελφους που δεν ε, μπορούσαν να παρευρεθούν. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές που θα, ε, θα ήθελα να τοποθετηθούν. Να είστε σίγουροι ότι έχετε το ενδιαφέρον μας παρά τη μικρή προσέλευση. Κυρία Μορβάη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτό την την εκπληκτική παρουσίαση που μας έδωσε πραγματικά άγνωστες μέχρι τώρα πληροφορίες και άγνωστα μέχρι τώρα συμπεράσματα. Εμείς, ε, εγώ εργάζομαι με θύματα βίας, ε, θύματα κακοποίησης, γυναίκες θύματα κακοποίησης. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι γίνεται με αυτά τα προγράμματα κατάρτισης για τη γυναική επιχειρηματικότητα. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να ε, στηρίξουμε τις ε, γυναίκες οι οποίες έχουν επιβιώσει από κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, ε, υπήρξαν θύματα πορνείας κτλ. Συνήθως χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος για να ξεπεραστούν οι τα αποτελέσματα της έμφυλης βίας. Πολλές γυναίκες χάνουν την αυτοπεποίθησή τους, την αυτοεκτίμησή τους. Πιστεύω λοιπόν πως ο καλύτερος τρόπος για να ε, βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες είναι να συνδυαστούν αυτά τα προγράμματα κατάρτισης πάνω στην επιχειρηματικότητα με άλλες ε, υπηρεσίες φροντίδας γυναικών που έχουν επιζήσει από κακοποίηση. Εσείς έχετε κάποια στοιχεία, κάποια εμπειρία σχετικά με το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα κατάρτισης επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες για γυναίκες θύματα βίας και κακοποίησης. Υπάρχει κάποιο νομικό ή κοινωνικό πλαίσιο που να στηρίζει τις γυναίκες. Υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες στην Ευρώπη και πώς μπορούμε να πληροφορηθούμε ε, για αυτές, πώς μπορούμε να μάθουμε περισσότερα Τώρα ε, σχετικά με την πρόεδρο μας είπατε ότι ζητήσατε, ζητάτε συγγνώμη για τη μικρή προσέλευση. 37 μέλη έχουμε στην Επιτροπή και είμαστε τρεις εδώ που έχουμε απομείνει μαζί με την πρόεδρο. Η αξιότιμη κυρία συνάδελφος είπε νωρίτερα ότι οι φασίστες και οι ρατσιστές δεν έρχονται σε συνεδριάσεις. Εγώ θέλω να πω σε όλους, ε, σε όλα αυτά τα πλήθη που μας παρακολουθούν από το ίντερνετ ότι δεν σημαίνει ότι το 95% που των μέλων της Επιτροπής είναι φασίστες, γιατί αν, το, αν κρίνεται από την προσέλευση και από αυτό που μας καταλογίζεται, τόσοι έχουμε μείνει. Δεν αρνούμε να απαντήσω, όχι πλάκα κάνω, είμαι ορισμένες φορές πολύ ειρωνική. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο τώρα στους ε, εμπειρογνώμονες ε, για να κάνουν ε, κάποια τελικά σχόλια. Ήσασταν ε, πραγματικά πολύ διεξοδικοί στις παρουσιάσεις σας. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Μουρβάη. Αν όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. for your question. First... Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Θα ήθελα να αφερθώ στο πρώτο κομμάτι της δηλώσής σας, δεν θέλω να πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Όντως ε, υπάρχουν ε, εμπειρίες που συνδέουν την προώθηση της επιχειρηματικότητας με δράσεις για συγκεκριμένες ομάδες γυναικών. Έχουμε τον Gold Rush, το κυνήγι του χρυσού που στη Γερμανία για 30 χρόνια υποστηρίζεται η μικροχρηματοδότηση. Ίσως ε, κάποια μέλη της Επιτροπής ε, γνωρίζουν την πρωτοβουλία, είναι μικρό το πρόγραμμα και η ομάδα στόχος είναι γυναίκες ε, που ε, έχουν υποστεί οικονομικοκοινωνική περιθωριοποίηση, μετανάστριες ως επιτοπλίστων ε, και το περιθώριο λάθος ε, αποτυχίας είναι 2 με 3%. Παρέχεται επίσης υποστήριξη, ε, βοήθεια για να οικοδομηθεί η αυτοπεποίθησή τους. Ο στόχος δεν είναι μόνο η σύσταση της επιχείρησης, μιλάμε για μια πέντα ετία και 72 νέες επιχειρήσεις, 240.000 ευρώ το κονδύλι. Ε, και ένα σύστημα για να αντιμετωπιστεί η περιθωριοποίηση, η καταπολέμηση της στόχης, ε, η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. Σωστά η Πρόεδρος μας έδωσε ε, και ένα παράδειγμα παραδοσιακών τομέων γυναικές επιχειρηματικότητας Έχουμε κι άλλο ένα παράδειγμα, 240.000, ή μάλλον αυτό το παράδειγμα 240.000 στο κονδύλι, 70 επιχειρήσεις. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ε, πάλι πενταετία στο Ηνωμένο Βασίλειο, 6 νέες επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν με 8 εκατομμύρια λίρες ε, στο τομέα ανάπτυξης ε, λογισμικών, δηλαδή καταλαβαίνετε υπάρχουν διαφορετικές προσδοκίες όπως σας έλεγα, διαφορετικά ταλέντα διαφορετικές δεξιότητες, όμως μέσα από αυτά τα δίκτυα, πέρα από τις οικονομικές δυνατότητες, όντως δίνουμε και δυνατότητες για, ε, κοινωνική, για κατοπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά, εύχομαι ό,τι καλύτερο και θα συναντηθούμε στην επόμενη μελέτη που θα ετοιμάσω. Δεν θα ήθελα να χαιρετήσω όλες τις παρούσες. Φτάνουμε στο τέλος. Θα τα πούμε αύριο στις 10 μετά από τη συνάντηση των συντονιστών και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι ψηφοφορίες.